przewodniczący! Panie i panowie, otwieram posiedzenie. Κυρίες και κύριοι, άρχεται η συνεδρίαση. Το πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξή μα προβλέπει δηλώσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τα συμπεράσματα της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 16 Σεπτεμβρίου 2010. Καλωσορίζουμε τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, κύριο Εργμάν Βαν Ρόμπεϊ. Καλωσορίζουμε τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το δίνουμε αμέσω το λόγο. Παρακαλώ κύριε πρόεδρε, έχετε το λόγο.